Δίνω το λόγο στην κυρία Μπόλς πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Λουσμονικών Υποθέσεων. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να εξηγήσω γιατί ζητάμε αναβολή του νομοθετικού ψηφίσματος, ούτω ώστε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, με την ενισχυμένη εντολή από την Ολομέλεια διεξήχθησαν δύο συζητήσεις επί του σημαντικότατου αυτού ζητήματος και είναι σαφέστατο ότι το να προσπαθήσουμε απλώς να έχουμε μια πλευρά να διαπραγματεύεται μόνη της και να λέει ότι δεν υπάρχει περιθώριο ελιγμών δεν είναι συναπόφαση, δεν είναι κάτι ικανοποιητικό εκτιμώ την υποστήριξη των συναδέλφων που στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα προς το Συμβούλιο στον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άντσες Μάλιστα. Εκ μέρου τη ηγήτρια κυρία Ελίζα Φεραίρα και μετά από συνεννόηση με του εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων και μετά τη γνώμη και τη Επιτροπή της Πρόεδρου της Επιτροπής και της Διάσκεψης Προέδρου προτείνω με βάση το άρθρο 57 παράγραφος 2 του κανονισμού να αναβληθεί η ψηφοφορία του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος. Γιατί αυτό που επιθυμούμε είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία ή δυνατόν στη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης με το Συμβούλιο. Γι' αυτό και ζητούμε από το Συμβούλιο να ακούσει το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας που πιστεύω ότι θα είναι σαφής και απερίφρεστη και να κινηθεί μετά από την επιστολή που θα λάβει από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με το θέμα αυτό. Καλώς. Άρα ζητούν από ό,τι φαίνεται την αναβολή του νομοθετικού ψηφίσματος, τόσο η πρόεδρος της Επιτροπής όσο και η συγγήτρια, δυνάμει του άρθρου 572. Ε, θα δούμε τώρα την ψηφοφορία όλων των τροπολογιών on block της αρμόδιας καθήλυνης επιτροπής, όμως η κυρία Φόρτ ζητάει το λόγο πρώτα. Συνάδελφοι, έχω δύο προφορικές τροπολογίες. Η μία είναι συντομότατη και οι δύο θέλουν να εξασφαλίσουν ότι τα προηγούμενα συμπεφωνημένα όσον αφορά την ενιαία αγορά, την έρευνα και ανάπτυξη, τι αρχέ που συμφωνήσαμε για την Τραπεζική Ένωση ε, γίνονται σεβαστά. Η πρώτη τροπολογία προσθέτει και μη συμμετέχοντες μετά από τη λέξη κάθε συμμετέχον ούτως ώστε κάθε χώρα να έχει λόγο όταν μια τράπεζα που έχει θηγατρική στη δικαιοδοσία της εμπλέκεται σε μια διαδικασία εκαθάρισης. Και οι δύο λοιπόν προτάσεις αφορούν το θέμα εκαθάρισης. Μάλιστα. Θέσατε, ακούσατε αγαπητοί συνάδελφοι την προφορική τροπολογία. Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις παρακαλώ να εγερθούν από τις θέσεις τους όσοι έχουν αντίρρηση. Χρειαζόμαστε άνω των 40 ορθίων. Νομίζω ότι είναι περισσότεροι. Λυπούμε κυρία Φόρτ. Επόμενη προφορική τροπολογία. Σας ακούμε. Thank you. Ευχαριστώ. Θα διαβάσω αυτή την τροπολογία αρκετά γρήγορα. Όπω φαντάζομαι θα έχουν αντίρρηση και για αυτήν οι συναδελφοί. Η τροπολογία είναι οι οποιοδήποτε ευθύνε τη Ένωση σε σχέση με μη συμβαλόμενε ευθύνε και που σχετίζονται με το κόστος και την επίδοση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού. Υπό οποιαδήποτε περίσταση δεν μπορεί να συνεπάγεται η αδίποτε οικονομική ευθύνη για τα κράτη-μέλη τα οποία δεν συμμετέχουν στο σύστημα. Τα μη συμμετέχοντα κράτη-μέλη. Τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη θα κάνουν διευθετήσεις ούτως ώστε τα μη συμμετέχοντα κράτη-μέλη να αποζημιώνονται πλήρω γρήγορα και με επιτόκιο με τόκο, σε σχέση με οποιαδήποτε ποσά που καταβάλλονται από τους ίδιους πόρους και όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για τους σκοπούς που αναφέρεται στην πρώτη υποπαράγραφο. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν σταματούμε την τραπεζική ε, ένωση, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρο πλέον που, ε, που βαρύνει το κόστος, ποιον βαρύνει το κόστος. Ε, ευχαριστώ. Καλώς, καλώς. Ευχαριστούμε. Απορρίπτονται και οι δύο προφορικέ τροπολογίε, δεν γίνεται δεκτή η ψήφισή του δηλαδή. Και περνάω στο αρχικό κείμενο τη Επιτροπή. Παρακαλώ, Γιάννη Γέρσεω. Κατά. Άποχες. Ένταξη. Παρακαλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τους μείωπες, γιατί εμένα μου ήταν πολύ ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 441 υπέρ. 141 κατά, 17 αποχές εγκρίνεται. Και τώρα, τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, παρακαλώ, διαναγερσός της χειρός, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα, το αίτημα δυνάμει του άρθρου 57 παράγραφος 2 για αναβολή της τελικής ψηφοφορίας, παρακαλώ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και σας ευχαριστώ. zunächst Herrn Enrique Iglesias, Generalsekretär. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εδώ να καλωσορίσω και τον Γενικό Γραμματέα της Αμεροϊβηρικής ε, ε, Διασκέψεως, ο οποίος μας επισκέπτεται επί τη ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής Eurolat. Καλώς ήρθατε. Και τώρα περνώ και πάλι στις ψηφοφορίες. ψήφισμα για τη χώρα καταγωγή και τον τρόπο προέλευση νοπού διατηρημένου σε απλή ψήξη ή κατεψυγμένου κρέατο χείρων, εγωπροβάτων και πουλερικών με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ψήφισμα για το σύστημα γενικευμένων δερμολογικών προτιμήσεων, ονομαστική και πάλι, παρακαλώ. Διαδικαστικό. Πρόεδρε. Δεν, ζητού, δεν απαιτούνταν ειδική πλειοψηφία για την προηγούμενη ψηφοφορία. Όχι για την επόμενη, λέει ο Πρόεδρος, για το σύστημα... Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων. Εδώ απαιτείται ειδική πλειοψηφία. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Απερίφθη. Και τώρα πιστοποιητικά εκπομπών 7α παράρφος 3 έχουμε αιτήματα από το EFD και το ECR και από τον κύριο Προτασίεβιτς και προτάσεις των βουλευτών για την πρόταση της Επιτροπής 1031-2010 για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την σημερινή ψηφοφορία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για τον το κανονισμό. Κύριε Πρόεδρε, με βάση το άρθρο 177-4 του κανονισμού, η ομάδα ε, υποβάλει επίσημο αίτημα ώστε να αναβληθεί η ψηφοφορία για την επόμενη Ολομέλεια. Γιατί αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και οδηγεί σε αύξηση των τιμών ενέργειας, του κόστου παραγωγής και του, της, ε, αυξάνει την ενεργεία. Άσχετα με την ιδεολογία του καθενός, Νομίζω ότι θα πρέπει να τηρήσουμε κάποιου κανόνε του παιχνιδιού και να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Αυτό ζητάει η FD. Θα πρέπει να αναλύσουμε πιο εντελεχώ την κατάσταση και μετά πιο εμπεριστατωμένα να λάβουμε μια απόφαση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ψηφοφορία γίνεται όπω ορίζει ο κανονισμός. Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται μόνο με τον κανονισμό. Ε, Επομένω μπορεί να μιλήσει κάποιο υπέρ, κάποιο κατά. Ποιο θέλει να ταχθεί υπέρ τη προτάσεω, κανεί κατά. Καλώ το ψηφίζουμε υπέρ τη αναβολή. Αναβολή υπέρ. Υπέρ τη αναβολή. Κατά. Απερίφθη. Ψηφίζουμε τώρα με ονομαστική ψηφοφορία. Κύριε Σπερώνη, δεν σας έδωσα τον λόγο. Δεν σας έδωσα τον λόγο κύριε Σπερώνη. Ζήτησα ποιος θέλει να μιλήσει νωρίτερα. Δεν ζητήσατε τον λόγο. Δεν είναι τσίρκο το κοινοβούλιο και ήδη ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Haben Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ψήφισμα σχετικό με την κατάσταση στην Ουκρανία. Υπάρχει κοινό ψήφισμα για την κατάσταση στην Ουκρανία. Ψηφίζουμε την πετετάρτη παράγραφο σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα το τρίτο κομμάτι της ψηφοφορίας. Αρχίζουμε. Ψήφισαν όλοι. <coughs> Πέρας. Εγκρίνεται. Μετά την 7η παράγραφο έχουμε τροπολογία 1 ονομαστικά. Προφορική τροπολογία, ο κύριο Σούλτ. Συνάδελφοι, το φω τη χθεσινής συζητήσεω και βλέποντα ξεκάθαρα τι γίνεται στην Ουκρανία, θα πρότεινα να πούμε σαφώ ότι είναι δικαίωμα του ουκρανικού λαού να αποφασίσει χωρί καμία διεθνή παρέμβαση για το μέλλον του. Και γι' αυτό προτείνω να αντικαταστήσουμε καταστήσουμε την τροπολογία 1 με την εξή διατύπωση και παραθέτω υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ουκρανικός λαός και μόνο αυτός θα πρέπει να αποφασίσει ελεύθερος από ξένη παρέμβαση για τη γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας και για το ποια διεθνή συμφωνία και κοινότητα θα πρέπει να προσχωρήσει η Ουκρανία και να προσθεθεί σαν μια νέα τελευταία φράση της παραγράφου 19. Όχι από ό,τι βλέπω. Προφορική λοιπόν τροπολογία, πρόσθετα στην υπαριθμό 1. Ποιος ψηφίσει ονομαστικά παρακαλώ, αρχίσει η προφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία και πάλι ονομαστικά παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Παράγραφος 14 στο αρχικό κείμενο, δύο τμήματα. Πρώτο παρακαλώ. Κατά. Κύριος Μπροκ, επί του κανονισμού. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μία παράληψη από πλευρά των ε, συντακτών της τροπολογίας αλλά και της σχετικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου ε, ε, έφερε ένα σφάλμα στην παράγραφο 14. Στη δεύτερη φράση πρέπει να γίνεται λόγος and the preparation, όχι introduction και την προετοιμασία μέτρων, όχι εισαγωγή. Προετοιμασία, preparation. Παρακαλώ να γίνει αυτή η διόρθωση. Ο Πρόεδρος, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι έχει γίνει η αποκατάσταση, μου λένε οι υπηρεσίες. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, στο πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και περνώ στο ψήφισμα για την κατάσταση στη Συρία. που έχει πολύ ψηλή θέση στο κατάλογο. Με πολλά ψηφίσματα, πιστεύω να βρείτε ο καθένα το ψήφισμα τη ομάδα σα. Κατάσταση στη Συρία. Κοινό ψήφισμα 6 ομάδων καταρχά. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε την τροπολογία 1, άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται το ψήφισμα στο σύνολό του παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κατάσταση στην Αίγυπτο τώρα. Πρόταση ψηφίσματος κοινή από έξι ομάδες. Υπάρχει μόνο δύο τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Παράγραφος 9 αρχικό τμήμα, αρχικό κείμενο δύο τμήματα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε για το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα στην παραγραφή 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία πρώτη υπέρ κατά αποχές πάλι δεν είναι σαφές. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την πρώτη τροπολογία. Αρχής ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απερίφθη ολόκληρο το ψήφισμα παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα το ψήφισμα για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας πράσινη καταρχάς πρώτα πρώτας ψηφίσματος της ομάδας των πρασίνων υπέρ κατά αποχές απερίφθη κοινό ψήφισμα πέντε ομάδων Παράγραφο 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά. Αποχέ απερίφθη, Παράγραφο 5, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχέ απερίφθη. Παράγραφο 6, αρχικό κείμενο, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνώ στο ψήφισμα για την έκθεση πρόοδου του 2013 για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 ονομαστικά Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. Εννέα στο αρχικό τμήμα, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε για το δεύτερο τμήμα της ένατης παραγράφου. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Η τροπολογία 2 έχει αποσύρθει ε, 29 αρχικό κειμένο πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 3 σε 2 τμήματα πρώτο υπέρ κατά απόχε εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, πάλι θα το δεύτερο τμήμα της, παρα, της τροπολογίας 3 αρχίζει η ψηφοφορία παρακαλώ ψήφισαν όλοι πέρας απερίφθη Επτά ονομαστικά. αρχής ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. Δεκαέξι ονομαστικά. Άρχισε ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη τη λογική σκέψη C, αρχικό κείμενο, σε δύο τμήματα, πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο υπέρ, κατά. Επαληθεύουμε για το δεύτερο τμήμα, αρχής ψηφοφορία. Είναι δύσκολο για μένα να παρακολουθήσω πώς ψηφίζουν οι πράσινοι, αν κανείς εδώ μπροστά δεν κάνει δεν δείχνει την ε, στάση της ομάδας. Ψηφίσαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και τώρα, ψήφισμα για... Κύριε Πόσλτ, του κανονισμού. Πρόεδρε, κατά, κατά εξαίρεση δεχθείτε μια μικρή παράβαση του κανονισμού. Κανείς δεν έχει προσφέρει τόσα στην Βοσνία Ερσεκοβίνη όσο η κυρία Πακ και νομίζω ότι πρέπει τώρα που ολοκληρώθηκε αυτή η ψηφοφορία να την ευχαριστήσουμε για τη δουλειά που έχει κάνει και την αφοσίωσή της 10 χρόνια τώρα. Κυρία Πακ, 600 περίπου άνθη σας ε, οφείλουμε σε ένα μεγάλο μπουκέτο. Και τώρα έχουμε την ψηφοφορία για την έκθεση πρώτου του 2013 για την πρώτη Οικοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Έχουμε την ε, πρόταση της Επιτροπή των Εξωτερικών, τροπολογία 4 υπέρ, κατά. Ε, δεν μπορώ να παρακολουθήσω πως κινούνται οι ομάδες Υπέρ. Υπέρ, τροπολογία 4. Κατά εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 22 αρχικό κείμενο δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 32 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά επαληθεύουμε μάλλον έχει απορριφθεί αλλά επαληθεύουμε αρχίζει η ψηφοφορία Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται παράγραφος 50 αρχικό τμήμα τα πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 3 έχει αποσυρθεί. Παράγραφο 51, αρχικό τμήμα, τόσο διατμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Τροπολογία, ε, κείμενο 58, αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα στην 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επαληθεύουμε το δεύτερο τμήμα στην παράγραφο 58 αρχικό κείμενο αρχίζει ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Αρχικό τμήμα κείμενο 59. Δύο τμήματα πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο ονομαστικά υπέρ. Αρχής προφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 ονομαστικά αρχίζει. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία πρώτη υπέρ, κατά αποχές στο σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά. Αρχής ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα προχωρούμε στο ψήφισμα για την έκθεση πρόοδο του 2013 για το Μαυροβούνιο και πάλι ψήφισμα της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων Τροπολογία πρώτη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαληθεύουμε. Αρχίζει. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη 3. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4-2 τμήματα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία Υπέρ. Κατά. Στενά τα περιθώρια. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 7 ονομαστικά άρχεται ψήφισαν όλοι πέρας το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται και περνάμε στο ψήφισμα για την εξάλληψη του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ψήφισμα της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών για την ισότητα των για των γυναικών. Πρώτη, τέταρτη παράγραφος, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη δέλτα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά ζητάτε επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της αιτιολογικής σκέψης ΔΕΛΤΑ, D αρχίζει η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρασε εγκρίνεται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και προχωρώ στο ψήφισμα που αφορά το πρόγραμμα ΝΑΙΑΔΕΣ 2, πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη εσωτερικής ναυσιπλοείας της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, πράγματος 3 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, ε, ονομαστικά, συγγνώμη, ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι, Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία πρώτη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Παράγραφος προ... ενδεκάτη στο αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη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 Καλή όρεξη και καλή επάνωδο. οποιο θέλει να λάβει μέρος στις επεξηγήσει ψήφου προφορικά παρακαλώ να μείνει στην αίθουσα. Οι λοιποί παρακαλώ ταχαίω και ησύχω να αποχωρήσουν. Ίσως θα χρειαστεί να καλέσω προσωπικά κάποιου συναδέλφου στην τάξη. Ξεκινώ με τι προφορικές τροπολογίες, καταρχάς για τα θέματα που δεν έγιναν εχθές, οι προφορικές ε, επεξηγήσεις ψήφου και μετά στα υπόλοιπα. Καταρχάς για την έκθεση Μπαχ.